Presidente. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να χαιρετήσω και το κοινό τόσο πολύ παρακολουθεί εδώ πέρα την συζήτησή μας. Η συνεδρία επαναλαμβάνεται. Τα συνοπτικά πρακτικά της Διεθνής συνεδρία και τα κείμενα που εγκρίθηκαν έχουν διανεμηθεί. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι τα συνοπτικά πρακτικά εγκρίνονται.